καθαρή ενέργεια με 30% όρο, δεσμευτικό όρο για το 2030 σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Η πρόταση είναι και ένα σοβαρό βήμα προς την επίτευξη των δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ολοκλήρωση της ε, Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης, Ένωσης και την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών διεθνώς. Η πρώτη ανταλλαγή απόψεων έγινε στις 23 Μαρτίου και σήμερα ο συγκεκριτή θα μας παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσής του. Αγαπητέ συνάδελφε κύριε Γκέρεκ, έχετε το λόγο. Σας ακούμε. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι. Το θέμα μας ε, είναι ήδη έτοιμο και η έκθεση έχει εκπονηθεί και μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες, οπότε μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στις προτάσεις που αφορούν το στόχο της ενεργειακής απόδοσης. Τώρα δεν θα σταθώ στο αν θα πρέπει να είναι 30% ο στόχος, 35% ή 40%. Το επίπεδο της φιλοδοξίας μας θα προκύψει από τις συζητήσεις με τις πολιτικές ομάδες. Εγώ πάντως προσωπικά θα προτιμούσα να έχουμε τον υψηλότερο δυνατό στόχο, γιατί θεωρώ ότι είναι εφικτός, επιτεύξιμος, αλλά είναι εφικτός ο στόχος αυτός μόνο και μόνο, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, γιατί δεν θα πρέπει να επικεντρώνεται μόνο στην ε, τελική ε, ενέργεια, αλλά να καλύπτει όλη την αλυσίδα από την πρωτογενή ενέργεια, να καλύπτει τη μεταφορά ενέργειας και το, την κατανάλωση ενέργειας από τον τελικό χρήστη, την τελική κατανάλωση και τη χρήση στην καταναλωτική αγορά. Είτε από τη βιομηχανία, είτε από τη γεωργία, είτε από, την, ε, από τα νοικοκυριά, τις κατοικίες, τον ε, κατασκευαστικό οικοδομικό κλάδο. Είναι λοιπόν ο στόχος εφικτός εφόσον καλύπτει όλη την αλυσίδα α, ε, της ενεργειακής απόδοσης από την πρωτογενή μέχρι την τελική ε, κατανάλωση. η γνωστή εποδός α, της έκθεσης είναι το θέμα της αξιοποίησιμης ενέργειας των ε, μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δηλαδή, οι, τα οι συντελεστές πρωτογενής, ε, πρωτογενούς ενέργειας, θα πρέπει να είναι ε, κοινά με τις προτινόμενες ε, τροπολογίες και να λαμβάνουν υπόψη και την έννοια της απόδοσης. Χρησιμοποιούνται για, την, για τον υπολογισμό της τελικής ενέργειας τη χρήση του, της τελικής ενέργειας για τον υπολογισμό της πρωτογενούς ενέργειας. Αυτό το σκοπό έχουν οι συντελεστές. Και εγώ πρότεινα κάτι που δεν περιλαμβάνει η προηγούμενη οδηγία του 2012. Γι' αυτό και ήταν δύσκολος ο υπολογισμός από την τελική ε, ενέργεια της πρωτογένους. Και θεωρώ ότι ήταν πολύ περιορισμένη η οδηγία του 2012. Γιατί Αλλιώς θα έχουμε μεγάλο περιορισμό στην πρωτογενή ενέργεια. Θα σας εξηγήσω τους λόγους. Ε, θα μπορούσαμε να μειώσουμε τις ε, εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου, να προστατεύσουμε το κλίμα, να διασφαλίσουμε και τους ενεργειακούς μας πόρους και να τους κρατήσουμε και για τις μελλοντικές γενιές, να μην εξαντληθούν. Και επίσης θα πρέπει οι εθνικές οικονομίες να αναπτύξουν την ανταγωνιστικότητά τους. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός βέβαια για τη χρήση ανανεώσιμων ποιών ενέργειας και αυτό, αυτή είναι η πρόθεση και της δικής μου έκθεσης. Αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός που σας ανέφερα, ότι και για την μετατροπή ανανεώσιμων ποιών ενέργειας σε αξιοποιήσιμη ενέργεια απαιτείται κάποια κατανάλωση ενέργειας. Δεν είναι 100% αποδοτική και αυτό το λέω στην έκθεση. Ε, και για να χρησιμοποιηθούν οι μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το ποσοστό τους εξαρτάται από το ενεργειακό μείγμα των χωρών μελών. Και ο στόχος της ενεργειακής απόδοσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με την αντικατάσταση ενεργειοβόρων τεχνολογιών και στην κατανάλωση και στην πρωτογενή ενέργεια με τη χρήση λιγότερο ενεργειοβόρων ε, ενεργειών ή την μεγαλύτερη πρόσβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και αυτή, αυτός είναι ένας ε, παράγοντας για μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση λαμβάνοντας υπόψη την έννοια της ορευτικής κατανάλωσης ενέργειας. Γιατί δεν θα πρέπει να συγχαίουμε την πρωτογενή με την τελική ενέργεια γιατί κάθε προϊόν έχει διαφορετικό τρόπο, ε, διαφορετικό τρόπο και μέθοδο ε, μετατροπής. Δεν μπορούμε να ε, συγκρίνουμε ε, μία λαμαρίνα με ένα εκλεπτισμένο όχημα. Έχουμε από τη μια πρωτογενή ενέργεια και από την άλλη τελική ενέργεια. Δεν θα πρέπει να τη συγκρίνουμε. Τώρα, για να υπολογίσουμε τις υποχρεώσεις των χωρών μελών για την περίοδο 2021-2030, ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ε, οικονομίες στην ε, σορευτική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας. Δεύτερον, θέλουμε μια ολιστική προσέγγιση όλων των οικονομικών κλάδων της, οικογένειας, της οικονομίας, ιδιαίτερα των ενεργειοβόρων και θα πρέπει να περιλάβουμε και τις μεταφορές. Επίσης, θα πρέπει να είμαστε ελαστικοί στην προσέγγιση των ε, κρατών μελών σε ό,τι αφορά την επιλογή τους ε, και τι θα διαλέξουν για να επιτύχουν την, ε, την ενεργειακή απόδοση. Και θα πρέπει η ενεργειακή απόδοση να καλύπτει όλους τους κρίκους αλυσίδα, την πρωτογενή ενέργεια, τη μετατροπή, τη μεταφορά, εδώ έχουμε τεράστια αποθέματα. Και θα πρέπει το κράτος μέλος να έχει επιλογή του τρόπου. Ε, με τον οποίο θα πραγματοποιήσει την ενεργειακή απόδοση. Και επίσης ε, η επιλογή του τρόπου επηρεάζει και το κόστος. Και έρχομαι στο κόστος, ιδιαίτερα στο επενδυτικό κόστος. Και να μην ξεχνούμε και την τελική καταναλωτική αγορά, τη, τη βιομηχανία, τα, νοικοκυρά, τα νοικοκυριά, τη στέγαση. Θα πρέπει και αυτά και αυτή τη φάση της τελικής κατανάλωσης να τη λάβουμε υπόψη. Σας ευχαριστώ. Έχουμε μια... σας συνάδελφός μας, κυρία Μπόσιουτ, που είναι και ε, αντιπρόεδρος της ΣΥΜΚΟ. Μάρκους Πίπερ, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αφού πρώτα καλωσόρισα την ε, συνάδελφό μας. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για την ε, σε βάθος ανάλυση και για την ε, επεξεργασία που έκανε στην πρόταση της Κομισιόν. Για τον υπολογισμό της πρωτογενούς ενέργειας υπάρχουν ορισμένα πράγματα και για τον συντελεστή αυτής της ενέργειας, οι στόχοι όπου, ε, και οι στόχοι επίσης όπου θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε. Ορισμένα πράγματα από αυτά που λέει τα βρίσκουμε πολύ ενδιαφέροντα και τα περιλαμβάνουμε και εμείς στον προβληματισμό μας, αλλά θέλω να σημειώσω επίσης ότι πρόκειται για επανεξέταση, review δεν πρόκειται για αναδιατύπωση ολόκληρης της οδηγίας. Ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να περιοριστούμε στα 3 έως 4 άρθρα που έχουν τεθεί ως αντικείμενο τη επανεξέταση και όχι όπως είπα νέα διατύπωση ολόκληρου του κειμένου της οδηγίας. Αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ ιδίω είναι να υπάρξει κάποια ευκαμψία, flexibility. Θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να δώσουμε αυστηρούς στόχους, χρειαζόμαστε ε, ρήτρα συγκυρίας, χρειαζόμαστε ενδεικτικούς στόχους και θεωρούμε επίσης ότι η συνεκτικότητα με το σύστημα ETS της εμπορίας των εκπομπών πρέπει να είναι ακόμα πιο συγκεκριμένη. Και εδώ θα αναπτύξουμε κάποιες ιδέες. Πρόκειται τέλος και για την διάρκεια που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να την ορίζει ως απεριόριστη εν τέλει. Θα βάλουμε εμείς σαφώς μια οροφή και θέλουμε να περιλάβουμε και τη δυνατότητα υπολογισμού και διαφόρων επενδύσεων, early actions δηλαδή, υπό την έννοια της ευκαμψίας υπέρ των χωρών μελών. Τελευταίο και επειδή συχνά αναφέρεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεση για την αποδοτική χρήση της ενέργειας, της οποίας ήμουν εισηγητής. Η έκθεση δεν ισχύει πλέον σε αυτές τις διαπραγματεύσεις διότι υπήρξε έκθεση η οποία ψηφίστηκε με πολύ μικρή πλειοψηφία. Υπερψήφισαν Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και ECR. Γι' αυτό αυτή η στόχη του 40% είναι απλώς ονειροπολίσεις. Και παρακαλώ και προς την κατεύθυνση του δημιουργούς διαλόγου να εμφανιστούμε ενωμένοι και όχι με κατακαιρματισμένη την θέση του Συμβουλίου, διότι στην περίπτωση αυτή το Συμβούλιο δεν πρόκειται να μας λάβει σοβαρά υπόψη. Ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα παίξουμε τον ρόλο μας, τον ρόλο μας εμείς, αλλά χρειαζόμαστε κάποια συνεργασία και από τις άλλες πλευρές. Πρόεδρος, ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Ακολουθεί. Κύριε Βανπόσιουτ, από τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη θα αναφερθώ στα πιο σημαντικά θέματα για τη δική μου πολιτική ομάδα, διότι για μας είναι σημαντικό να λάβουμε ως στόχο τα ενδεικτικά 30%. Την στόχευση δηλαδή και για την μείωση του δικτύου του άνθρακος. Οι δε χώρες μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να επενδύσουν εκεί όπου διαβλέπουν μεγαλύτερο δυναμικό. Μπορούν να είναι ανανεώσιμε πηγές ενέργειας, μπορεί να είναι αποδοτική χρήση της ενέργειας και ούτω καθεξής. Τώρα για την πρωτογενή και την τελική ενέργεια θεωρούμε ότι είναι σημαντικό οι χώρες μέλη να λάβουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν το σύστημα το οποίο χρησιμοποίησαν πάντοτε. Ορισμένες χώρες μέλη βασίζονται ιδίω στην πρωτογενή ενέργεια, άλλες στην τελική αυτό σημαίνει ότι οι χώρες μέλη για μας πρέπει να έχουν δυνατότητα επιλογής σε ό,τι αφορά το άρθρο 7. Για τις ετήσιες μειώσεις κατά 1,5%. Εδώ συμφωνούμε με το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο δεν προτείνει 1,4%. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό το έτος 2027 να γίνει μια αξιολόγηση διότι όπως είπα και πριν θα έχουμε πια ήδη συλλέξει τους ε, καρπούς που είναι στα χαμηλότερα κραδιά. Θα έχουμε τελειώσει με αυτά τότε και τα πράγματα θα γίνουν ακριβότερα. Και θα χρειαστεί να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος πλέον στην αποδοτική χρήση ενέργειας. Και ίσως μπορούμε τότε να στοχεύσουμε περισσότερο σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να μειώσουμε το δεξιό του άνθρακος. Τέλος, για το παράδειγμα 5. Εκεί είναι σημαντικό να διατηρηθεί η ευκαμψία υπέρ των χωρών μελών για την επίτευξη των στόχων. Θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε ορισμένα πράγματα και να υπονομεύσουμε την ίδια τη δική μας νομοθεσία, διότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία στην περίπτωση αυτή δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Πρέπει να συζητήσουμε θέματα όπως επισήμανση της ενέργειας, για να πείσουμε και τον καταναλωτή ότι μπορεί να αγοράσει ένα ας πούμε ψυγείο ή άλλη ηλεκτρική συσκευή με καλύτερη αποδοτικότητα από ό,τι πριν. Χρειάζεται λοιπόν όλα αυτά να συνυπολογιστούν στους στόχους. Η κυρία Αγγέλικα Μίλνερ που αντικαθιστά τον κύριο Γκερμπράντι, ο οποίο είναι πάλι και ο ε, των φιλελευθέρων. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ. Αντικαθιστώ τον Χερμπερτιάννη και Μπράντι αλλά και του συναδέλφου μου από την ομάδα μα. Ε, συνάδελφοι, πριν από ένα χρόνο η ε, πρόταση για την ενεργειακή αποδοτικότητα συνδυάζεται με την Ενεργειακή Ένωση για την Ευρώπη. Ε, Στου φιλελευθέρου έχουμε τι εξή απόψει. Πρέπει να αγωνιστούμε για την ασφάλεια τη εφοδοσία, την απαλλαγή από τον άνθρακα, την ε, μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικέ τιμέ ενέργεια. Δύο χρόνια αργότερα, μετά την πρώτη πρόταση, οι υποθέσει που είχαμε κάνει στην υποβολή τη ε, ισχύουν. Πρέπει να δούμε τι συνέπειε των κλιματικών αλλαγών που λένε και εντείνονται, γίνονται ορατότερε καθημερινά και να δούμε την ε, παγκόσμια κούρσα για την καθαρή ενέργεια. Η Κίνα έχει ε, επενδύσει 300 δις ευρώ για να γίνει πρωταγωνίστρια στον χώρο αυτό και ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να αγωνίζεται με όλα του τα μέσα κατά τη συμφωνία των Παρισίων, όμως ο ιδιωτικός τομέας καταλαβαίνει ότι το οικονομικό μέλλον ε, έχει να κάνει με την καθαρή ενέργεια. Καθαρή ενέργεια που θα είναι φτηνότερη και ανταγωνιστική, Δεν σας αρέσει όχι. Γι' αυτό καλωσορίζω την δεσμέτρων καθαρή ενέργεια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλου του Ευρωπαίου. Το συνολικό αυτό πακέτο θέλει να δημιουργήσει μια νέα αγορά, ενισχύοντα ε, την ενέργεια και επιτρέποντα τη μετάβαση προ ανανεώσιμε πηγέ και τη χρήση του. Ωστόσο, εάν θέλουμε η ενεργειακή μετάβαση να πετύχει, πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Εάν θέλουμε να συμμορφωνόμαστε με του ε, στόχου τη Συμφωνία του Παρισίων το 2015, πρέπει να είμαστε φιλοδοξότεροι και να δράσουμε άμεσα. Για να πετύχουμε του στόχου των κλιματικών αλλαγών, η ενεργειακή αποδοτικότητα πρέπει να υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Εξοικονομώντα ενέργεια, θα μειώσουμε τι εκπομπέ. Θα έχουμε καθαρότερου ουρανού και υγιέστερο περιβάλλον. Επιπλέον, θα μειωθεί το κόστο τη ενέργεια και για τι επιχειρήσει και για του πολίτε. Θα γίνουμε λιγότερο εξαρτώμενοι από τι εισαγωγέ ενέργεια. Και τελευταίο, αλλά εξίσου σοβαρό, θα δημιουργήσουμε θέσει απασχόληση που τόσο πολύ χρειάζεται όλη η Ευρώπη. Βεβαίω, οι επιχειρήσει θα καταλάβουν ότι αν θέλουν να επιβιώσουν μακροπρόθεσμα πρέπει να είναι προστατευμένε ω προ τι ελλείψει ενέργεια. Θα πρέπει τα προγράμματα ενεργειακή αποδοτικότητα να επιτρόψουν ιδιωτικέ επενδύσει μέσω όμω δεσμευτική νομοθεσία. Θέλουμε επίση επενδυτική βεβαιότητα με μια μακροπρόθεσμη θεώρηση. Γι' αυτό να αυξηθεί ο στόχο μα το 40% σε δεσμευτικό επίπεδο για όλα τα κράτη-μέλη. Για να κάνουν ε, οι χώρε όλε τι προσπάθειε που χρειάζονται και να επιτύχουμε αυτού του φιλόδοξου στόχου. Πρέπει να υπάρξουν λοιπόν εθνικοί δεσμευτικοί στόχοι. Για να πετύχει ενεργειακή μετάβαση πρέπει να εργαστούμε μαζί σε όλα τα επίπεδα. Να συνεργαστούμε με τι επιχειρήσει, τι εθνικέ κυβερνήσει, τι τοπικέ αρχέ με τι πόλει και του πολίτε. Για να ολοκληρώσω, συνάδελφοι, είναι πολύ ψηλό το διακύβευμα. Αν θέλουμε ε, καθαρή, ασφαλή ενέργεια, πρέπει να δράσουμε όλοι μαζί από κοινού. Ελπίζω ειλικρινώ να συμφωνήσουμε σε μια φιλόδοξη ε, θέση του Ευρωπαϊκού, Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που να επιτρέπει χειροπιαστέ μακροπρόθεσμε δράσει. Οι Ευρωπαίοι περιμένουν από εμά και αξίζουν τη δράση μα. Ελπίζω να έχουμε καλή ε, συνεργασία στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία μου. Ο κύριος Γιάβορ από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον ε, εισηγητή για, την, ε, για το σχέδιο έκθεσή του και πιστεύω ότι μπορούμε να εργαστούμε επικοδομητικά για να πετύχουμε μία οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα που να είναι φιλόδοξη τουλάχιστον από την πλευρά του Κοινοβουλίου, και να δημιουργήσουμε ένα σταθερό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Είμαι και ο στην Επιτροπή ΕΝΒΗ και ήδη είχαμε την πρώτη συνάντηση σκιωδών στην Επιτροπή μα και βλέπω να υπάρχουν κάποιε κοινέ μέρημνε μεταξύ των ε, πολιτικών ομάδων, κάτι που αποτελεί μια καλή βάση για τη συνέχεια τη συζήτηση και την εξετάση του θέματο. Σε γενικέ γραμμέ, Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε πόσο σημαντική είναι η οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα προκειμένου να εφαρμόσουμε τη Συμφωνία των Παρισίων. Κάτι απαραίτητο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να διατηρήσουμε αμύωτη τη φιλοδοξία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είχαμε συμφωνήσει και προηγουμένω ε, για το 40%. Το είχαμε πει και σε περασμένε περιστάσει. Στι συζητήσει με το Συμβούλιο Βλέπω να υπάρχει μια θετική τάση στις εξελίξεις και στις συζητήσεις μας, αλλά δεν φτάνει. Χρειάζεται σταθερή δέσμευση από το Κοινοβούλιο για τα θέματα της ενεργειακής αποδοτικότητας και το σχετικό φάκελο και για να παραμένει σε ορθή πορεία η ε, διαδικασία της οδηγίας για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Πιστεύω να υπάρχουν κάποια, ε, ότι υπάρχουν κάποια σημεία σύγκλησης κάποιο κοινό έδαφος για να εργαστούμε επί του θέματος και να κατονομάσω μερικά. Πρέπει να κάνουμε τους ιστούς συσχετισμούς με τα υπάρχοντα νομοθετήματα, τον οικολογικό σχεδιασμό και την οδηγία του, αλλά και το σύστημα ανταλλαγή εκπομπών, το ETS, δεδομένων και των διαθεσμικών διαπραγματεύσεων για την αναθεώρησή του. Καθώς και άλλα τμήματα τη ε, οδηγία για την καθαρή ενέργεια, το EPDD, τα ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, την χρηματοδότηση και ούτω καθεξής. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε και εδώ θα συμφωνήσουμε με τον κύριο Πίπερ ότι μιλάμε για αναθεώρηση της οδηγίας. Οπότε αντί να την ε, αναδιαρθρώσουμε πλήρως, ας ε, διατηρήσουμε την γενική διάρθρωση, κλείνοντας λόγω χάρη τα κενά στο άρθρο 7, για να εξαιρεθούν από τη βασική γραμμή οι μεταφορές στα κράτη-μέλη, λόγω χάρη. Επίσης θα πρέπει να γίνουν κάποιες προσαρμογές για την ε, μακροπρόθεσμη προοπτική μας και τους στόχους μείωσης των εκπομπών για την Ευρωπαϊκή Ένωση με ορίζοντα το 2050. Ε, για την ιδιωτική και κρατική επενδυτικότητα στην ιδιωτική, στις ιδιωτικές επενδύσεις χρειάζεται σταθερότητα στο μακροοικονομικό περιβάλλον, ασφάλεια και ε, δυνατότητες για να χρηματοδοτηθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα, ενώ οι, οι κρατικές επενδύσεις πρέπει να επικεντρωθούν στους ευάλωτους καταναλωτές. Χρειάζεται και κρατική χρηματοδότηση παρόλα αυτά για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Και τελευταίο, πρέπει να αναφέρω ότι είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε και στην, στο κατασκευαστικό, στον τομέα των κτηρίων και τα δημόσια κτίρια. Χρειάζονται επιπλέον οικονομίες στον ε, τομέα αυτό. Με τα κτίρια μηδενικής ε, ενεργειακής κατανάλωσης βάσει των προτύπων που υπάρχουν και πρέπει να επικεντρωθούμε και σε αυτό το στόχο. Ευχαριστούμε πολύ, συνάδελφε, για τις παρατηρήσεις σας. Επόμενος ομιλητής είναι ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ήτρε, ο κύριος Κόχλιτσεκ, που εκπροσωπεί την ΚΟΕ. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έχω αρκετές παρατηρήσεις. Όταν μιλούμε για την ενεργειακή απόδοση, θα πρέπει να είμαστε σαφείς ως προς τον επιδιωκόμενο στόχο. Αν βάλουμε στόχο το 30%, είναι ρεαλιστικός στόχος και θα πρέπει να καλύπτει όλους τους ε, οικονομικούς κλάδους συμπεριλαμβανομένων και των μεταφορών. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι τα κτίρια έχουν ε, μακρά διάρκεια ζωής. Πολλά κτίρια, ιδιαίτερα ε, στα κέντρα των πόλων, είναι διατηρηταία. Και για τέτοια κτίρια είναι πολύ ε, δύσκολο να βάλουμε, ε, να τα θωρακίσουμε, να κάνουμε μια θερμική αναβάθμιση, δηλαδή να βάλουμε επένδυση που θα εξασφαλίζει θερμομόνωση. Επίσης υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ βορρά και νότου των κλιματικών συνθήκων και αυτό επηρεάζει την ενεργειακή απόδοση. Όλα τα βήματα που θα πραγματοποιήσουμε για την ολοποίηση αυτού του στόχου θα είναι διαφορετικά από χώρα σε χώρα. Επίσης, ε, ποια ενέργεια θα ληφθεί υπόψη, η πρωτογενής ή η τελική. Εγώ δεν θα ήθελα να επικεντρωθούμε μόνο στην πρωτογενή ενέργεια και στους αντίστοιχους πόρους, γιατί αυτό θα μας φέρει πάλι πίσω στην ε, αιωλική ενέργεια, όταν ε, οι αεροστρόβιλοι είχαν μηδενική ισροή. Το ίδιο και η φωτοβολταϊκή ενέργεια. Και τα γνωρίζω αυτά. Άσχετα μιλάμε για βαριά μέταλλα, χαλκό ή αποσύνθεση των στοιχείων για τους α, ε, στρόβιλους. Όλα αυτά απαιτούν μεγάλη ενέργεια σε επίπεδο ισρών. Μεγάλη πρωτογενή ενέργεια. Και αν εξετάσουμε το θέμα της παραγωγής χαλκού, από άποψη απόδοσης ενεργειακής ε, είναι πολύ χειρότερος ο χαλκός και η παραγωγή χαλκού από άλλους ε, ενεργειακούς πόρους. Γι' αυτό λέω να αφήσουμε κατά μέρου ε, από τον υπολογισμό δηλαδή την πρωτογενή ενέργεια ή τουλάχιστον να αρχίσουμε να τη συμπεριλάβουμε σε μεταγενέστερα στάδια. Και φυσικά εξαρτώνται όλα αυτά από το ενεργειακό μείγμα και τους, πόρους που, τους ενεργειακούς πόρους που χρησιμοποιούμε για να υπολογίσουμε την πρωτογενή ενέργεια. Ευχαριστώ. Παίρναμε τώρα μετά τους και οδησίγητες στους λοιπούς εισηγητές. Ο κύριος Μαχτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τον εισηγητή μας τον κύριο Γκέρεκ για τις προσπάθειές του και το έργο του. Ε, λυπάμαι πάντως που θα εκφράσω κάπως διστάμενη άποψη. Παρόλο που ανήκουμε στην ίδια πολιτική ομάδα, δεν συμφωνούμε σε όλα. Και θα παρουσιάσω τις διαφωνίες μας εδώ. Εγώ θεωρώ ότι σήμερα οι κλιματικές αλλαγές, είτε είναι κανείς υπέρ είτε κατά, είναι πραγματικότητα. Και δεν το λέω αυτό επειδή σήμερα έχουμε 33 βαθμούς στις Βρυξέλλες. Όλοι συμφωνούμε ότι θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε τον ενεργειακό μας ανεφοδιασμό και όλοι συμφωνούμε να τηρήσουμε τη συμφωνία της COP21 και να έχουμε μια φιλόδοξη πολιτική ώστε να μην υπερβούμε τους δύο βαθμούς ε, σε ό,τι αφορά τη θέρμανση του πλανήτη. Σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας εκπομπών, είμαι από αυτούς που ε, έχουν εκνευριστεί και απογοητευτεί γιατί δεν ήμασταν αρκετά φιλόδοξοι και δεν θεωρώ ότι θα καταφέρουμε με την αναθεώρηση να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Τέλος πάντων, επειδή είμαι δημοκράτης, υποκλίνομαι στην πλειοψηφία. Πάντως, ε, καλό θα ήταν να εξασφαλίσουμε μη τι άλλο αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές και τους προσανατολισμούς. Μην ξεχνάτε ότι ο στόχος μας μέχρι το 2050 είναι μια βιομηχανία με μηδενικές εκπομπές άθρακα. Αυτό είναι ο στόχο για το 2050. Ωραία τα λόγια βέβαια, αλλά θα πρέπει να τα εφαρμόσουμε, να περάσουμε, ε, να περάσουμε στα έργα. Και έχουμε και το πακέτο για την καθαρή ενέργεια για όλου του Ευρωπαίου, που έχει ως βασικό άξονα και ως πρωταρχική προτεραιότητα την ενεργειακή απόδοση. Από αυτή την άποψη, η τη της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση θα αποτελέσει στοιχείο κλειδί του συνολικού πακέτου και ακρογωνιαίος λίθος της Ενεργειακής Ένωσης. Και εδώ έχω κάποιες διαφωνίες και λυπάμαι ειλικρινά που δεν μπορώ να ασθενιστώ όλους τους στόχους του εισηγητού συμφωνώ να καλύψουμε και την παραγωγή, την ε, μετάδοση, τη μεταφορά και την κατανάλωση, όλους τους κρίκους δηλαδή της ε, παραγωγής ενέργειας και της ε, κατανάλωσης, αλλά από, διαβάζοντας την έκθεση βλέπω ότι επικεντρώνεται στους ανάντι Και έτσι περιορίζουμε τη δυνατότητα των κρατών μελών να, τηρήσουν τους στόχους χρησιμοποιώντας την καλύτερη εξοικονόμηση στην παραγωγή ενέργειας και να επηρεάσει ταυτόχρονα και την ε, καταναλωτική συμπεριφορά. Κατά τη γνώμη μου, έτσι δεν θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε το στόχο μας της καταπολέμησης της ενεργειακής ένδυας. Εδώ ο εισηγητής προσπαθεί να καλύψει αυτούς ε, του παρόχου ενέργεια που θεωρεί ότι θα μειώσουν τι ε, τιμέ των ενεργειακών προϊόντων και άρα θα μειωθούν οι λογαριασμοί ενέργεια. Βέβαια, αυτό είναι μια υπόθεση. Δεν είναι δεδομένο ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Και επίση ε, ε, δεν υλοποιεί το στόχο τη οδηγία. Και μάλιστα έτσι ώστε δημιουργήσουμε μια επισφαλή κατάσταση και μεγαλύτερη ενεργειακή ένδυα. Και μάλιστα θα έχουμε δύο χαμένους εδώ στην περίπτωση αυτή ε, τους ε, καταναλωτές και το κλίμα και μόνο ένα κερδισμένο τον παραγωγό της ενέργειας. Επίσης, ε, υπάρχει στενή σχέση μεταξύ, ε, την έκθεση, της ενέργειας, του περιβάλλοντος για του κόστους. Δεν συμφωνώ. Θα πρέπει να σχετίσουμε δύο παράγοντες. Την ενεργειακή απόδυση με το βασικό εργαλείο της αποσύνδεσης. Εμείς, οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες, χρόνια ολόκληρα επισημέναμε ότι θα πρέπει να διεκδικήσουμε το στόχο του 40% ενεργειακή απόδοση και μάλιστα ως δεσμευτικό στόχο. Θα δούμε μετά ποια βάση θα χρησιμοποιήσουμε για τον υπολογισμό. Αν θα είναι κριτήριο αναφορά το 2005 ή το 2007. Δεν μας ενδιαφέρει το έτος αναφοράς. Το σημαντικό είναι αν με τη συγκεκριμένη οδηγία θα θέσουμε φιλόδοξους στόχους ώστε να υλοποιήσουμε και τις φιλοδοξίες της συμφωνίας του κλίματος. Το ETS, το σύστημα ε, εμπορίας εκπομπών, είναι να μην βλάψει αυτούς που ήδη το εφαρμόζουν. Ουσιαστικά, τους ρηπαίνοντες απαλλάσσουμε από την καταβολή των ε, ε, τελών για τη ρήπαση που επιφέρουν. Ουσιαστικά, τους παραγωγούς ενέργειας, λοιπόν, ωφελούμε με την έκθεση αυτή και ευδυνούμε και όχι τον καταναλωτή το κλίμα. Για όλους αυτούς τους λόγους θα καταθέσω και τροπολογίες. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Ελπίζω ότι είχατε την ευκαιρία να τοποθετηθείτε πλήρω, έτσι είναι. Κύριε Μάρτεν, ευχαριστώ. Θαυμάσια λοιπόν. Η κυρία Στέρφερ, που είναι και ε, διευθύντρια στην Γενική Διεύθυνση Ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά, καθώς, ε, κύριε πρόεδρε πάνω, καθώς και τον καθηγητή κύριο Γκέρεκ για την προσέγγιση που έχει επιλέξει και ιδίως όσον αφορά εξοικονομήσεις ενέργειας που να αποδίδουν και στο κόστος παντού όπου είναι δυνατόν αυτό σε όλη την αλυσίδα. Επίσης για τον φιλόδοξο στόχο σαφώς άνω του 27% η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότισε, πρότεινε ως δεσμευτικό στόχο τα 30% για να υπάρχει αυτή η προβλεψιμότητα υπέρ των επενδυτών, ασφάλεια για τις επενδύσεις, να γίνουν δηλαδή επενδύσεις στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και κυρίως και στα κτίρια. Ο στόχος θα βασιστεί σε υπολογισμό μάλλον, θα της ε, εξοικονόμηση θα βασιστεί σε ένα έτος αναφοράς. Το βασικό άρθρο είναι το άρθρο 7 για την αναθεώρηση της οδηγίας. Και θα γίνει μάλιστα Δευτέρα ένα σημαντικό Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας και εκεί θα, συζητηθεί και το επίπεδο του άρθρου 7. Χρειάζεται λοιπόν να διατηρηθεί ο φιλόδοξο στόχο που έχουμε στα χέρια μα ήδη και αυτό περιλαμβάνεται ακριβώ στο αναθεωρημένο κείμενο αποδοτική χρήση τη ενέργεια. Θέλουμε λοιπόν το ίδιο να διατηρηθεί το ίδιο επίπεδο 2018, 19, 20 και τουλάχιστον μέχρι το 2030. Άρα η αντίποτε απόπειρα αποδυνάμωση του άρθρου 7 δεν είναι καλή. Και θεωρούμε πολύ καλό και καλοδεχόμαστε αυτό που προτείνει ο κύριος Γκέρεκ, δηλαδή λιγότερες ευκαμψίες σε πρόορες δράσεις που δεν θα συνυπολογίζονται στη νέα περίοδο ή ο υπολογισμό τη πρωτογενούς ενέργειας που κατανώνεται στις ε, μεταφορές. Θέλω να τονίσω επίσης ότι η ο υπολογισμο τη πρωτογενους ενεργειας που καταναλωνεται στις μεταφορες θελω να τονισω επισης οτι η εκθεση μας βοηθεί και για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, ώστε να ωφεληθούν οι καταναλωτές από την, ε, μετα, ε, με τον μετασχηματισμό ενέργειας. Πρέπει να διευκρινίσουμε ίσως ένα ή ζητήματα διότι η προτινόμενη διαγραφή της βασικής αρχής της προσθετικότητας είναι δύσκολη, διότι αυτή η προσθετικότητα θα διασφαλίσει οι εξοικονομήσεις αυτές να γίνονται επιπροσθέτως των όσων συμβαίνουν χάρη σε άλλες πολιτικές ή νομοθετικές ενέργειες της Ένωσης. Άρα θα είναι πρόσθετα μέτρα αυτά. Και αυτό θα πρέπει να απηχείται στο κείμενο της αναθεώρησης όπως το πράττει τώρα. Το δεύτερο τονίστηκε και από άλλους, είναι η έμφαση στον τομέα μετασχηματισμού της ενέργειας. Αυτό δεν θα πρέπει να γίνει σε βάρος των προσπαθειών που γίνονται από την άποψη της ζήτησης της ενέργειας, από την πλευρά δηλαδή της ζήτησης της ενέργειας. Θέλουμε βέβαια να δώσουμε βάρος στην κατανάλωση γενού ενέργειας, νομίζουμε όμως και είναι σημαντικό. Στο άρθρο 3 Εάν βασιστούμε μονάχα στην κατανάλωση πρωτογενούς ενέργεια, αυτό δεν επαρκεί. Χρειάζεται να έχουμε στόχο και για την τελική ενέργεια και θα πρέπει να διατηρηθεί ο στόχο αυτό, ώστε να απηχεί όλε τι επιτυχημένε πολιτικέ που έχουμε ήδη. Το ίδιο ισχύει για το άρθρο 7. Θα πρέπει να διατηρήσει την στόχευσή του για την κατανάλωση τελική ενέργεια. Εκφράζω τι σκέψει αυτέ και με τι σκέψει αυτέ εκφράζω και την ικανοποίησή μα για το περιεχόμενο της εκθέσεως του καθηγητού Γκέρεκ και βεβαίως θα δώσουμε κάθε δυνατή υποστήριξη στην Επιτροπή σας. Ευχαριστώ. Είναι μέρος της επιστημονικής επανάστασης αυτή η προσέγγιση του κ. Γκέρεκ. Άντα ήρθε η ώρα μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης να ξαναλάβεις το λόγο για να κάνεις μια ανακεφαλαίωση και να αντιλήσει και κάποια συμπεράσματα. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Άκουσα με μεγάλη χαρά τις παρατηρήσεις των συναδέλφων και τις σημείωσα. Νομίζω ότι είμαστε σε θέση να καταλήξουμε σε συνένεση. Και ε, ενδεχόμενες διαφωνίες δεν προκύπτουν από ε, το διαχωρισμό της πολιτικής ιδεολογίας. Δεν είναι ε, διαφορά, οι διαφορές μεταξύ των πολιτικών ομάδων, αλλά περισσότερο μεταξύ των χωρών, των πιο εύφορων και των ε, πιο φτωχών χωρών. Γιατί διαφορετικά προσεγγίζουν την ε, αξιοποίηση, την εκμετάλλευση της αγοράς ή τον περιορισμό. και όπως είπε ο κύριος Μαρτάν, δεν αγνοούμε την αγορά, αντίθετα το λαμβάνουμε υπόψη, αλλά λέμε ας, αφήσουμε, στα κράτη-μέλη την ε, διακριτική ευχαίρεια να διαλέξουν με τι θα ασχοληθούν. Ας ε, διαφυλάξουμε την ευελιξία, αυτή την ελαστικότητα στην αλυσίδα ροής ενέργειας. Φυσικά υπάρχει και το τελικό σκέλος, η τελική ενέργεια, αλλά εδώ θα ήθελα από την αρχή να πω το εξή. Οι χώρες που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, διότι ε, Τρει-τέσσερι φορές λιγότερο από άλλε. και μάλιστα η πατρίδα μου και η Ρουμανία και πολλές χώρες, ε, για να μην πω όλες, κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης που είναι σύμφωνες με την, ε, με την έκθεσή μου, Χώρε αυτές που έχουν πολύ χαμηλότερη παραγωγή ενέργειας προσεγγίζουν πολύ διαφορετικά αυτά τα θέματα. Εκεί το 40% περιορισμό τη ενεργειακή κατανάλωση είναι για αυτούς, ισοδυναμία για αυτούς με μείωση του ακαθάριστου χώρου προϊόντος. Κάτι που δεν ισχύει για το Λουξεμβούργο ή τη Σουηδία. Εκεί η κατανάλωση ενέργειας είναι τετραπλάσια. Ούτε συμφωνώ με εκείνους που λένε «Α, η οικονομία είναι ανεξάρτητη από την ενέργεια και σήμερα έχουμε μια κατάσταση όπου μπορούμε να έχουμε ένα ιδιαίτερο περπέτου μόμπιλε. Όχι, δεν μπορεί να λειτουργήσει η οικονομία χωρίς ενέργεια. Επίσης, δεν α, αυξάνονται με παρόμοιο τρόπο τα ΑΕΠ ή μειών, μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας. Υπάρχει ένα συνδυασμό μεταξύ τους. Δεν είναι αυτόματο ότι το ένα αυξάνεται και το άλλο ε, μειώνεται. Επίσης, το τελικό, θα, θα είναι η τελική ενέργεια. Μα η τελική ενέργεια ούτως ή άλλως στη στατιστική θα ληφθεί, θα ληφθεί υπόψη. Και το είτε τη συμπεριλάβουμε εμείς στον υπολογισμό είτε όχι, ούτως ή άλλως θα ληφθεί υπόψη ε, η τελική ενέργεια για να κριθεί το πώς επηρέασε η αύξηση των τιμών το γενικό πληθυσμό. Η υπόθεση όμως ότι ε, κάθε ενάμιση χρόνο θα μειώνουμε την ε, προσφορά ενέργειας στην αγορά, ενώ οι μικρότερες χώρες, ούτως, οι φτωχότερες χώρες ούτως ή άλλως δεν έχουν αρκετή ενέργεια. Αυτό πραγματικά ισοδυναμεί με βαρβαρότητα. Μια τέτοια προσέγγιση είναι βάναυση. Οπότε δεν θα πρέπει να το ε, εξετάζουμε ξεχωριστά. Θα πρέπει να βλέπουμε την αξιοποίηση της πρωτογενούς ενέργειας κυρίως, γιατί η πρωτογενής ενέργεια είναι αυτή που εκπέμπει ε, διοξίδιο του άνθρακα. Η τελική ενέργεια είναι καθαρή. Και αν θέλουμε να απαντήσουμε και να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις του Παρισιού, την πρωτογενή ενέργεια θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, όχι την τελική. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Πάντως χαίρομαι που και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχτηκε κάποιες προτάσεις μου. Φυσικά λάθη γίνονται και από νομική άποψη. Εγώ δεν είμαι νομομαθής, αλλά είναι καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ρυθμίσει το νομικό ζήτημα και να προσαρμόσει τα τεχνικά μέτρα στις ε, νομικές διατάξεις, ώστε να υπάρχει συνοχή της τελευταίας πρότασης και της αναθεώρησης οδηγίας με τα προηγούμενα ε, με το προηγούμενο νομοθετικό έργο. Έχω εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα επιτύχει τη νομική ευθυγράμμιση των διαφορών νομοθετικών πράξεων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, αγαπητέ συνάδελφε. Για τις τροπολογίες έχετε προθεσμία μέχρι τις 28 Ιουνίου του 2017, μέχρι την επόμενη Τετάρτη δηλαδή ουσιαστικά, έχετε τη δυνατότητα να καταθέσετε τροπολογίες. Λίγο χρόνο έχετε, μόλις 6 μέρες. Περνάμε τώρα στο δεύτερο θέμα του απογεύματο, στην πρόθεση τη χρήση ενέργεια από ανανεώσιμε πηγέ. Χωσέ Μπλακό Λόπε, ο εισηγητή. Η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρήση ενέργεια από ανανεώσιμε πηγέ είναι ένα από τα α, ε, κλειδιά, τα βασικότερα σημεία του πακέτου για την καθαρή ενέργεια. Και λέει δεσμευτική ευρωπαϊκή στόχη 27% για το μερίδιο της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην μεικτή γενική ε, κατανάλωση μέχρι το 2030. Και μάλιστα μερικές ε, προτάσεις ε, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Περιβάλλοντος, όπως αποφάσισε το Μάιο η διάσκεψη των Πρόεδρων. Έγινε ήδη μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων στις 23 Μαΐου, η Μαρτίων μάλλον, συγγνώμη, και σήμερα ο εισηγητής μας, ο κύριος Χωσέ Μπλάνκο Λόπες, θα μας παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσής του. Κύριε Σιγητά, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τη γραμματεία της Επιτροπής και κυρίως την Ελβίρα και την γραμματεία του Κοινοβουλίου, καθώς και τους ε, εμπειρογνώμονες της Επιτροπής ε, και τους ε, συμβούλους, καθώς και του, το, τους υπαλλήλους της Σοσιαλιστικής Ομάδας για τη μεγάλη βοήθεια που μου πρόσφεραν. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε ε, τη μαρτυρία της Προέδρου των νησιών Μάρσαλ στην Ολομέλεια του Στρασβούργου. Και μπορεί ο πρόεδρο των ΗΠΑ να αφιβάλλει για τι κλιματικέ αλλαγέ, αλλά τα νησιά Μάρσαλ δεν έχουν καμία απολύτω αμφιβολία οι κλιματικές αλλαγές είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια απτή πραγματικότητα και αδιαφυσβήτητη. Και ο Ντόναλτ Τραμπ αντί να στηριχθεί σε επιστημονικές αποδείξεις ε, αμφισβητεί αυτές τις επιστημονικές έρευνες και τα συμπεράσματα και αποσύρει τη χώρα του από την ε, Συμφωνία των Παρισίων. Χαρακτηρίστε τη συμπεριφορά του όπως θέλετε. Ανευθυνότητα, ασυνέπεια, θράσος, όλα αυτά ισχύουν. Και εγωισμός υπερβολικός εγωισμός, γιατί η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση. Και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει αυτή η ενέργεια να μα αποθαρρύνει στον αγώνα καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών. Θα πρέπει αντίθετα να εντείνουμε τι φιλοδοξίε μα και τι δράσει μα. Και μάλιστα τα συμπεράσματα του G7 ενισχύοντας τις δεσμεύσει των παγκόσμιων εταίρων είναι ένα πολύ θετικό βήμα. Το ίδιο και το ότι ε, κρατήσαμε την ενότητα και την ακεραιότητά μας ε, απέναντι στην, στην ε, συμπεριφορά του Ντόναλτ Τραμπ και διατρανώσαμε την προσήλωσή μας στο, στη Συμφωνία του Παρισιού. Εμείς είμαστε στην καλή πλευρά της ιστορίας, σίγουρα, αλλά όχι αρκετά. Το είδαμε και στη συζήτηση της Ολομέλες, ώστε ο αρνητισμός του Τραμπ είναι η μοναδική απειλή στις κλιματικές αλλαγές, αλλά άλλες απειλές είναι ε, απλώς αγαθές προθέσεις και δεσμεύσεις μόνο στα λόγια, χωρίς να περνάμε στα έργα, χωρίς να διορθώνουμε ε, τα μέτρα για το πακέτο των, της καθαρής ενέργειας. Γιατί όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να γίνει πιο φιλόδοξη η σχετική οδηγία. Η της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απάδει από τους στόχους των Παρισίων για απεξάρτηση από τον άνθρακα μέχρι το 2050 και να μην υπερβούμε την αύξηση τη θερμοκρασία του πλανήτη κατά δύο βαθμού, μειώνοντα το διοξείδιο του άνθρακα. Αν δεν χαράξουμε ενεργειακέ και κλιματικέ πολιτικέ ε, συμβατέ με το, τη Συμφωνία του Παρισιού, είναι σαν να απαρνούμαστε του στόχου μα. Μέχρι στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν υπόδειγμα, παράδειγμα προ για τον κόσμο και είμαστε σε καλή θέση για να απαλλάξουμε την οικονομία μα από θρακούχε εκπομπέ. Τώρα περισσότερο από ποτέ θα πρέπει να δείξουμε πυγμή, αποφασιστικότητα, να γίνουμε υπόδειγμα προ και να πρωτοστατήσουμε στην ενεργειακή μετάβαση. Μάλιστα, το κόστο των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια έχει μειωθεί. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή τη μείωση για να έχουμε φτηνή ενέργεια, για να εξασφαλίσουμε ενεργειακή αυτάρκεια και να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα. Και δεν αρκεί ο στόχο του 27% για τις ΑΠΕ. Ούτως ή άλλως, χωρίς να κουνήσουμε τα δαχτυλάκια μας όταν πετυχαίναμε. Προτείνω λοιπόν να ανεβάσουμε αυτό το ποσοστό στο 35% για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ναι, μεν είναι φιλόδοξος ο στόχος, αλλά είναι και λογικός και ρεαλιστικός και εφικτός. Επίση, προτείνω δεσμευτικού στόχου για τα κράτη-μέλη. Κάτι τέτοιο θα εξασφαλίσει ασφάλεια δικαίου και είναι αναφυσβήτητο μήνυμα υπέρ των ΑΠΕ. Ταυτόχρονα ε, τονώνει την, ε, ε τις επενδύσεις ε, και θα συμβάλλει στη μείωση του κόστους. Θα πρέπει όμως ταυτόχρονα να προβλέψουμε κάποια κριτήρια για τα συστήματα στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να ξεπεράσουμε την αφησιμία. Γι' αυτό και προτείνω συγκεκριμένα κριτήρια για τα κράτη-μέλη, για, τον, για τη διοργάνωση διαγωνισμών και να λάβουν υπόψη για την μετάβασή τους περιβαλλοντικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες θα πρέπει φυσικά να ενισχύσουμε και την ρυθμιστική και κανονιστική ασφάλεια. Μάλιστα, οι μέχρι τώρα πολιτικέ μα για τι ΑΠΕ δημιούργησαν αβεβαιότητα στου επενδυτέ, ε, θέτω σε αναφιβόλο την υλοποίηση των στόχων του 2020 και βλάπτοντα τη βιομηχανία. Η ανάπτυξη λοιπόν τη ασφάλεια δικαίου θα έχει θεμελιώδη σημασία για να εξασφαλίσουμε και να κάνουμε πιο φθηνέ επενδύσει στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Γι' αυτό ενισχύουμε το άρθρο 6 για να διασκεδάσουμε τις αμφιβολίες και τις ανησυχίες και να εξασφαλίσουμε μέλλον στις τωρινές επενδύσεις. Επίσης, ακόμη και αρνητικά προγράμματα που έχουν απορριφθεί θα πρέπει να, λάβουν κάποια αποζημίωση. Θα πρέπει και ο καταναλωτής να συμβάλλει με την αυτοπαραγωγή για ίδια κατανάλωση. Και επίσης θα πρέπει να αρθούν τα διοικητικά εμπόδια, ώστε ε, ενέργεια που μένει στο δίκτυο να μην χρεώνεται. Νομίζω κάτι τέτοιο είναι πολύ δίκαιο για τους καταναλωτές. Σε ό,τι αφορά την θέρμαση και την ψήξη, αλλά και σε ό,τι αφορά τις μεταφορές, ο τομέας αυτός αντιπροσωπεύει το 30% της κατανάλωσης ενέργειας και κυριαρχείται από τα παράγοντα του πετρελαίου και τα ορεκτά καύσιμα. Θα πρέπει λοιπόν να θεσπίσουμε μέτρα που πραγματικά θα ευθυγραμμίζεται με το δρόμο που άνοιξε η Συμφωνία του Παρισιού. Γι' αυτό όμως χρειάζεται μεγαλύτερη φιλοδοξία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην οδηγία της. Επίσης, ο πρόεδρος Γιούνκερ στον οδικό χάρτη για την θετία του τόνισε ότι θα πρέπει να αυξήσουμε το μερίδιο των ΑΠΕ στην Ήπειρό μας. Συμφωνώ μαζί του και πιστεύω ακράδαντα ότι είναι μεγάλο το δυναμικό της οικολογικής ανάπτυξης αυτών των ΑΠΕ. Και θεωρώ ότι έτσι θα μπορέσουμε να κατακτήσουμε την πρώτη θέση παγκοσμίω στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Πιστεύω με κάθε ταπεινότητα ότι οι προτάσει αυτέ με ε, συνεπή, εφικτό και αποτελεσματικό τρόπο θα μα βοηθήσουν να υλοποιήσουμε του στόχου μα. Σα ευχαριστούμε πολύ, συνάδελφοι. Και τώρα οι σκιώδει εισηγητέ. Ο κύριο Σον Κέλλη, εκ μέρου του ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Μπλάνκο Λόπες για την ε, εισήγησή του, για το σύνταξη της έκθεσης και την ξεκάθαρη ένδειξη ότι θέλει να έχουμε μια ομαλή συνεργασία για το θέμα αυτό. Πράγμα που δείχνει και η πράσινη γραβάτα του. Ναι, Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να συγκεράσουμε τις διαφορετικές απόψεις. Πολλά από τα σημεία που θίξατε με βρίσκουν σύμφωνο. Τα προγράμματα στήριξη των ανεώσιμων στο μέλλον ε, μας βρίσκουν σύμφωνους, όπως και αυτά που προτείνατε για το όλο σύστημα. Πρέπει να δώσουμε μια μακροπρόθεσμη ε, ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα για τους επενδυτές για να υπάρξει μια ομαλή αγορά. Οι προτάσεις του εισηγητή λοιπόν για την διοργάνωση διαβουλεύσεων και οι ειδικοί κανόνες για τις προμήθειες καθώς και τα, οι προϋποθέσεις για να μπορεί κανείς να συμμετάσχει είναι σωστά στοιχεία. Κατά την άποψή μου πρέπει να βρωθεί σωστή ισορροπία μεταξύ του πολιτικού κόστους που θα πρέπει να είναι χαμηλό, των ε, τιμών ενέργειας που θα πρέπει επίσης να είναι ε, λογικές και την επίτευξη των στόχων για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να οργανώσει ανοιχτού ε, διαγωνισμού και προμήθειε. Όμω θα, χρειαστούν και προγράμματα στήριξη σε κάποιε περιπτώσει. Η χρήση νέων τεχνολογιών, η χρήση τοπικών ενεργειακών πόρων, η σταθερότητα μακροπρόθεσμα στα καύσιμα και ούτω καθεξής. Θα πρέπει αυτά να αναφέρονται ρητό στο κείμενο τα προγράμματα στήριξη και το άνοιγμά του σε διασυνοριακή συμμετοχή. Είναι ένα βήμα που καλωσορίζουμε στην πρόταση τη Επιτροπή. Όμω, αν, αν το εννοούμε σοβαρά και θέλουμε να εφαρμόσουμε την Ενιακή Ένωση, πρέπει να υπάρχουν σωστοί κανόνε. Και να είμαστε και προσεκτικοί για το πώ θα το, ε, θα το διατυπώσουμε. Ο κύριο Μπλάνκο Λόπε λέει να είμαστε φιλόδοξοι και να υπάρχει ένα μεγάλο άνοιγμα τη αγορά. Όμω, να φροντίσουμε, ε, να προσέξουμε σε αυτό το νέο πεδίο που θα ανοίξει μπροστά μας και να είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα στην πράξη. Μην προκύψουν καταστάσεις όπου κάποια έργα θα επιλέγονται βάσει του που είναι χαμηλότερο το κόστος και οι φόροι και όχι με το που υπάρχουν μεγαλύτερες με ανάγκες οι πόροι. Θα δημιουργηθούν μία συμφόρηση και αυτό πρέπει να προσέξουμε. Ένα άλλο στοιχείο που καλωσορίζω είναι η επιθυμία του ε, εισηγητή να ενισχυθεί η βεβαιότητα των επενδυτών. Είναι σημαντικό αυτό και στην αγορά των ανανεώσιμων πηγών και καλωσορίζω τις προτάσεις του κυρίου Λόπες. Η αναδιαναμητική ε, διάσταση είναι σημαντική, αρκεί να υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις για την αυτοκατανάλωση και ιδίως για το κοινοτικό μοντέλο. Είναι σημαντικό να μην υπάρχουν ε, τέλη εφόσον δεν είναι αποτελεσματική επιβολή τους. Σε αυτό θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε με τον εισηγητή. Παρόλα αυτά πρέπει να γίνει μια διευκρίνηση. Το, το κείμενο θα πρέπει να διασφαλίζει την αρχή ότι κάθε χρήστης του δικτύου δεν θα ε, υποφελείται από θετική διακριτική μεταχείριση. Το σύστημα πρέπει να είναι δίκαιο, να επιτρέπει τη συμμετοχή όλων και να μην ε, παίρνει το κόστος από κάποιους χρήστες για να το μεταφέρει σε άλλους, ώστε να είναι και μακροπρόθεσμα βιωσιμότερο. Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη στα πλαίσια αυτής της οδηγίας, αλλά είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να βρούμε το σωστό σημείο ισορροπίας. Για την θέρμανση και την, ε, τον κλιματισμό μπορούμε να συζητήσουμε πολύ. Ε, στην θέρμανση πρέπει να απαλλαγούμε από τον άνθρακα μακροπρόθεσμα και να φτάσουμε στο στόχο του 2%, τον δεσμευτικό στόχο που πρότεινε ο εισηγητή. Αλλά αυτό ίσω να είναι υπερβολικά φιλόδοξο. Θα πρέπει να υπάρξει ευελιξία για τα κράτη-μέλη, ώστε ο στόχο για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργειας να επιτευχθεί με τρόπο ε, αποτελεσματικό και ω προς το κόστος. Ε, τόσο υψηλό δεσμευτικό στόχο ίσω να είναι υπερβολικό, αλλά αυτό θα το συζητήσουμε και ίσω να συμφωνήσουμε. Και μετά για τι μεταφορέ. Ο εισηγητή έκανε κάποιε ενδιαφέρουσε προτάσει, ιδίω με τον πολλαπλασιαστή για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα. Είναι θετικό αυτό, ε, δεδομένων των γοργών εξελίξεων στις τεχνολογίες ε, των ηλεκτροκινήτων για τα καύσιμα και μετά την πρώτη φάση της σταδιακής, μετάρι με... σταδιακής κατάργησης και μείωσης θα περάσουμε μοιραία προς τα ΒΙΒΙ και νομίζω ότι ε, κακώς δεν εξετάζουμε αυτό το θέμα εμείς αλλά η Επιτροπή ΕΝΒΗ θα έπρεπε να έχουμε και εμείς εδώ ένα λέγην. πάντως πέραν των δεσμευτικών στόχων πρέπει να έχουμε ισχυρά κίνητρα ώστε να μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα αυτά θα παίξουν ρόλο στην απαλλαγή από τον άνθρακα του όλου τομέα των μεταφορών. Τώρα για τον συνολικό στόχο του 27%. Ο Επίτροπος Κανιέται είπε το πρωί εδώ ότι η Επιτροπή θα ξαναδεί το στόχο αυτό υπό το φως των ε, σημερινών εξελίξεων και βάσει των νέων αποδεκτικών στοιχείων. Προτού λοιπόν ε, κάνουμε σχόλιο γι' αυτό, επιφυλασσόμαστε. Ευχαριστώ για την υπομονή σας, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Ιδιαίτερη περίπτωση σήμερα ιδιαίτερη περίστασα. Ε, ελεύθερος χρόνος αγόρευσης. Είδατε τι καλό σπίτι είμαι. Για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές, ο κύριος Τοσενόφσκι, που αντικαθιστά τον κύριο Χένκελ, τον αντιπρόεδρό μας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Συγγνώμη εκ μέρους του κυρίου Χένκελ, ο οποίος έχει υπερβολικά πολλές λιμένες υποχρεώσεις και δουλειές σήμερα, οπότε μου ζήτησε να σα διαβάσω το κείμενο του ως σκιώδου εισηγητού. Ο κύριος Χένκελ είναι της άποψης ότι πρέπει να επιτύχουμε κατά μέσο όρο τον στόχο του 30% μέχρι το 2030. Το ψήφισμα του Κοινοβουλίου του 2014 ε, ακριβώς αυτό λέει και προτείνει. Επιπλέον ο κύριος Χένκελ βάσει των όσων προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προβλέπει και δεν θεωρεί ότι τα κρατημέλη θα εγκρίνουν δεσμευτικούς στόχους. Βεβαίω πρέπει να αποσταλεί κάποιο πολιτικό μήνυμα προς τους επενδυτές ώστε οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επιτυχία τους να βασιστούν σε αγορές όπως τις προτείνει η Επιτροπή. Εάν έχουμε μια προσέγγιση ολιστική, σφαιρική και λάβουμε υπόψη και άλλες ε, περιπτώσεις όπως την ελεύθερη εμπορία του ηλεκτρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ισχυρή περιφερειακή συνεργασία, την απελευθέρωση της αγοράς του ηλεκτρισμού ε, της ηλεκτρικής ενέργειας μακροπρόθεσμα, τότε ίσως πετύχουμε καλύτερες τιμές για όλους τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Ο κύριος Χένκελ πιστεύει ότι στη μεταβατική περίοδο προ την απαλλαγή από τον άνθρακα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα βιοκαύσιμα και για τι μεταφορέ. Σε πολλά κράτη-μέλη ήδη υπάρχουν σχετικοί φιλόδοξοι στόχοι. Όμω, σε αυτή τη μεταβατική φάση, τα κριτήρια ε, βιωσιμότητα πρέπει να είναι ακλόνητα και να υπάρχει ένα σύστημα που να ε, μην επιτρέπει την αποψήλωση τρίτων χωρών προκειμένου να πετύχουμε εμεί του στόχου μα εδώ. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε. Από τους φιλελευθέρους, και πάλι η κυρία Μλίναρ, η οποία ε, αντικαθιστά τον κύριο Φέντερλε που είναι συντονιστής για την ομάδα των φιλελευθέρων. Έχετε το λόγο, κυρία μου. Ευχαριστώ πολύ. Ο Φέντερικ Φέντερλε δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα το απόγευμα, ζητάει λοιπόν συγγνώμη και καταρχάς θέλει να ευχαριστήσει τον εισηγητή για το σχέδιο έκθεσης θα είναι ένα καλό σημείο αφετηρίας για τις συζητήσεις μας η μετάβαση προς μια πρασινότερη και απαλλαγμένη επάνθρακα οικονομία δεν είναι απλώς προϋπόθεση για την περιβαλλοντική μας ευρωστία, αλλά είναι απαραίτητη για να υπάρξουν νέες καινοτόμες θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ένωση να παράγει περισσότερη ενέργεια από εσωτερικού ευρωπαϊκούς πόρους. Οι επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας από νέους εγχώριους πόρους θα μας επιτρέψουν να έχουμε και μεγαλύτερη ασφάλεια στην τροφοδοσία. Ε, επιπλέον, η νέα οδηγία για τι ανανεώσιμες πηγές είναι σημαντική όχι μόνο γιατί θα μπορεί να θέσει φιλόδοξου στόχου, αλλά είναι και μέρο ε, των ρυθμιστικών θεμελίων για τι επιχειρήσει και για να υπάρξουν οι επενδύσει που χρειαζόμαστε για να πετύχουμε του στόχου μα. Και ε, εν τέλει, μακροπρόθεσμα να βεβαιωθούμε ότι φτάνουμε του στόχου τη Συμφωνία των Παρισίων. Ε, Ενδεχομένω, ο συνολικό στόχο μπορεί να είναι μεγαλύτερο από την αρχική πρόταση τη Κομισιόν. υπάρχουν γοργέ εξελίξει στι τεχνολογία την τελευταία χρονιά και ταυτόχρονα μια μείωση του κόστου. Ε, θέλουμε πρωταγωνιστικό ρόλο για τα θέματα τη ενέργεια και των κλιματικών αλλαγών. Έχουμε τώρα μια τεράστια ευκαιρία εμεί να φανούμε ε, παγκόσμια πρώτη ε, στην προσπάθεια να απαλλαγούμε από τον άνθρακα στην οικονομία μα. Ε, η οδηγία αυτή είναι ένα σημαντικό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να οδεύσουμε προ αυτό το στόχο μπορούμε να δημιουργήσουμε το κατάλληλο πλαίσιο με κίνητρα ε, τις ε, ε, επενδύσεις που να βασίζονται στις ανάγκες και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνη μεταξύ των επενδυτών. Είναι ζωτική σημασία η οδηγία αυτή να μην γίνεται αντιληπτή ως κάτι που θα παρεμποδίσει την ανάπτυξη, την πρόοδο της αγοράς στις ανανεώσιμε πηγές ενέργειας και να δράξουμε την ευκαιρία αυτή για να προσπαθήσουμε να εκφράσουμε τις σωστές αρχές ώστε να μπορέσουμε στην επερχόμενη αναθεώρηση να αποφύγουμε να ξανανοίξουμε συζήτηση για τα ίδια θέματα. Ο φάκελο αυτό δεν θα είναι απλό, χρειάζεται υψηλό επίπεδο συντονισμού, επειδή υπάρχουν προεκτάσει και σε άλλα θέματα τη ενέργεια, αλλά και λόγω τη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ τη δική μα Επιτροπή με την Επιτροπή ΕΝΒΗ. Ιδίω όταν γίνεται λόγο για φιλοδοξίε στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, πρέπει να ξανασκεφτούμε θέματα που θα κοιτάξει και η Επιτροπή ΕΜΒΗ. Λόγω χάρη, πώ θα χρησιμοποιήσουμε του εσωτερικού μα πόρου, του εγχώριου πόρου και τι κανόνε θα θεσπίσουμε για να γίνει αυτό, καθώ θα υπάρχει άμεσο αντικτυπώ για το εφικτό, για το κατά πόσο θα επιτύχουμε του στόχου για τι ανανεώσιμε πηγέ. Αυτά όλα πρέπει να τα σκεφτούμε στι εργασίε μα. Δεν θα είναι απλό. Χρειάζεται πολλή δουλειά, αλλά ε, εύχομαι να είμαστε επικοδομητικοί στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για να φτάσουμε στο επίπεδο των φιλοδοξιών μας και να έχουμε ένα καλό ρυθμιστικό περιβάλλον για τις επενδύσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, κυρία Μλίνερ. Ο κύριος Κλωτούρμας τώρα από τους Πράσινους. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τον κύριο Μπλάνκο Λόπες, γιατί όντω ήταν ε, πολύ αξιόλογο το μέχρι τώρα έργο του και θα αποτελέσει εξαιρετική βάση για τη συζήτηση. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις. Μ' άρεσε πολύ προσέγγιση του Σον Κέλλη να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Θα αναπτύξω περαιτέρω αυτό το θέμα. Για τους στόχους τώρα, το πρώτο μείζον ζήτημα. Να αντιληφθούμε ότι το κόστος των ΑΠΕ έχει πέσει κατακόρυφα και για τις ε, ανεμογεννήτριες, τις επίγες τις υπεράκτιες, ε, τις θαλάσσιες, τις Οπότε, ακόμη και ο Διεθνής Οργανισμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ε, έχει προτείνει ε, ε, ένα στόχο 33% ως προς την αποτελεσματικότητα σε σχέση με το κόστος των ΑΠΕ. σε σχέση με τα, τις εκπομπές του 2013-2014. Και μάλιστα τις προάλλες είχαμε ένα πρόγευμα εργασίας με εμπειρογνώμονες από πολλά μέρη της Ευρώπης και ίσως ε, ε, στη διάρκεια του καλοκαιριού θα αποσαφινιστούν ε, τα πορίσματα των επιμέρους μελετών και το Σεπτέμβριο θα έχουμε μια πιο εμπεριστατωμένη συζήτηση για το ακριβές ποσοστό, το κατάλληλο ποσοστό για το μερίδιο των ΑΠΕ. Πάντως, η ΑΠΕ είναι πολύ σημαντική η επένδυση που σημαίνει κεφαλαϊκό κόστος και γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε βεβαιότητα για τους επενδυτές χωρίς αναδρομικές αλλαγές. Η αναδρομική ισχύση των αλλαγών είναι ο εφιάλτης κάθε επενδυτή. Επίσης θα πρέπει να απαλείψουμε και άλλους κινδύνους για τους επενδυτές και γι' αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε τα άρθρα 4 και 5 του κοινού εγχειριδίου κανόνων. Θέλουμε ε, διαγωνισμούς ε, ειδικού για τη τεχνολογία με κειμενόμενα σε επιδοτήσει. Οπότε αν αυξηθεί ή βελτιωθεί καλύτερα, αν βελτιωθεί η τιμή του ε, του άνθρακα, να ληφθεί υπόψη σε ένα κειμενόμενο ποσό. Και αν μέσα σε πέντε χρόνια βελτιωθεί η τιμή στη αγορά ε, ε, με μείωση του λόγου κόστους ε, αποδοτικότητας, αυτόματα να μειώνεται το ποσό, το, το τέλος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ώστε για τους επενδυτές να έχουν μια μακροπρόθεσμη προοπτική 15-20-25 χρόνων. Αυτό χρειάζονται. Και ένα άλλο θέμα που θα πρέπει να αποφύγουμε, ένα άλλο κίνδυνο είναι τα δίκτυα. Ε, μας ενδιαφέρει η πρόσβαση, πρόσβαση κατά προτεραιότητα και κανόνες για τον περιορισμό. Και επίσης ε, το διασυνοριακό χαρακτήρα. Η Ιρλανδία έχει καταπληκτικό απόθεμα ελληνική ενέργεια. Αν όμω κλείσει, ε, υπάρχουν σύνορα, θα χρειαστούμε καλώδια για να πάνε στη Γαλλία ε, τα, ε, η ενέργεια. Το ίδιο πρόβλημα θα έχει και η Ισπανία, η Πορτογαλία. Οπότε το θέμα του δικτύου θα πρέπει να μας απασχολήσει. Ε, σε ό,τι αφορά τι μεταφορές και τα, τη θέρμανση και την ψήξη, θα πρέπει και στη και ψήξη και στις μεταφορές αυξήσουμε το ποσοστό των ΑΠΕ. Θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία, γιατί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε βιομάζα, αλλά η βιομάζα ε, είναι ανταγωνιστική με τα χημικά προϊόντα, με τις ζωτροφές, τα τρόφιμα, ε, περιορίζεται από την βιοπικιλότητα. Υπάρχει ένα όριο στη βιομάζα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και θα πρέπει να είναι διαθέσιμη όποτε τη χρειαζόμαστε. Σε ό,τι αφορά τα βιοκαύσιμα, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, γρήγορη τουλάχιστον εναλλακτική για τα αεροπλάνα. Καλύτερα λοιπόν να, να επικεντρώσουμε το θέμα το, ε, να επικεντρωθούμε στο θέμα των βιοκαυσίμων ε, στα ε, οχήματα όπου υπάρχει η εναλλακτική της ηλεκτροκίνησης και ας αφήσουμε προς το παρόν τα αεροπλάνα και να δούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε διάφορες πηγές ανανεώσιμων ε, ενεργειακών μέσων. Να λάβουμε υπόψη και τον ηλεκτρισμό και το ίδιο να κάνουμε και τη θέρμανση και την ψήξη. Γεωθερμική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια επίσης ε, είναι σημαντικές ή ε, αντιλίες θερμότητας και αυτές ε, είναι λύσεις που μπορούμε να διερευνήσουμε. Χρειαζόμαστε όμως χρόνο για όλα αυτά και τέλος χρηματοδότηση όπως είπα και την προηγούμενη φορά. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα κυρίω για τι χώρε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Έχουμε υψηλότερο κεφαλαϊκό κόστο στην Πολωνία, Ρουμανία ή Βουλγαρία σε σχέση με τη Γερμανία και τη Γαλλία. Οπότε τα ίδια, οι ίδιοι ηλιακοί συλλέκτες, οι ίδιες ανεμογεννήτριες στην Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία κοστίζουν περισσότερο ακριβώς γιατί είναι πιο επικίνδυνη επένδυση για την αγορά. Ό,τι έκανε η Παγκόσμια Δράπεζα για το Μαρόκο θα πρέπει να το εφαρμόσουμε και στην Ευρώπη. Να αφαιρέσουμε τον κίνδυνο από τα επικίνδυνα τέτοια ε, σχέδια. Και όταν ένα σχέδιο θεωρείται κοινωνικού ενδιαφέροντος, να χρηματοδοτείται από κοινοτικά κονδύλια, ώστε να μειωθεί το κόστος, το κεφαλαιακό στις χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Και επίσης να εμπλέξουμε και τους πολίτες στο παιχνίδι. Γιατί όχι ένα ταμείο που και συνεταιριστικέ οργανώσεις να έχουν πρόσβαση σε φθηνότερο κεφάλαιο. Πολύ ευχαρίστω να συζητήσουμε πιο διεξοδικά κάποια άλλη φορά όλε αυτές τι ιδέες. Ε, ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Κλοντ. Έξι λεπτά το τονίζω αυτό διότι θέλω να σου δείξω πόσο τυχερός είσαι. Ευχαριστώ για την κοινοδορία σου, Πρόεδρε. Ζανονάτο, ο επόμενος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με τη γενική διάρθρωση του θέματος που μας έχει προτείνει ο εισηγητής και τον ευχαριστώ για την άριστη δουλειά του. Το κείμενο είναι πληρέστατο και μάλιστα και προηγμένο σε σχέση με τις ε, περιορισμένες φιλοδοξίες της ε, πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι φιλόδοξο. Δύο σημεία λοιπόν και ε, αργότερα επιφυλάσσομαι να κάνω λεπτομερέστερα σχόλια. Πρώτον, για το στόχο του 35% που προτείνεται τον εισηγητή. Συμφωνώ Πρέπει να ανακτήσουμε και να εδραιώσουμε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παγκοσμίω, διότι σήμερα σε όλες τις ε, περιπτώσεις γύρω μας με τις εξελίξεις, όπως με την ε, Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, βλέπουμε να δημιουργούνται τρεγμοί και ανησυχίες. Φοβάμαι όμως, όπως και ο Μπλάνκο, ότι ο στόχος του 35% στο, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να είναι τελικό σημείο προορισμός μας, όχι το σημείο αφετηρίας. Ως προς αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις, ώστε αυτό να είναι το σημείο όπου θα καταλήξουμε, όχι το σημείο από το οποίο θα ξεκινάμε. Να το ε, συζητήσουμε λοιπόν αυτό το σημείο αφετηρίας, εάν θέλουμε μετά από διεξοδικές διαπραγματεύσεις να έχουμε ελάχιστο στόχο 35%. Δεν φαντάζομαι ότι θα είναι απλό. Ίσως τότε το ποσοστό να πρέπει να αυξηθεί για την πρώτη φάση των διαπραγματεύσεων. Η δεύτερη μου παρατήρηση έχει να κάνει με ένα πρόβλημα που αφορά λίγο πολύ όλες τις εκθέσει, ε, οι οποίες κάποιες φορές επικαλύπτουν διαφορετικούς τομείς. Οπότε όταν κάποιες φορές θέματα έχουν άλλες προεκτάσεις είναι δύσκολο να μην αναλάβουν περισσότερες από μία επιτροπές. Ε, εδώ υπάρχει πρόβλημα λοιπόν με την ένταξη των ανανεώσιμων στις αγορές και εντός αυτού το πρόβλημα του ορισμού της προτεραιότητας πρόσβασης και ε, αποστολής. Είναι άλλη νομοθετική πρωτοβουλία αυτό, το γνωρίζω καλά, αλλά ταυτόχρονα και εκεί ανησυχώ για τον ενδεχόμενο κίνδυνο, δεν μπορούμε να μην δούμε το θέμα των ανεώσιμων πηγών ενέργειας χωρίς να ε, κοιτάξουμε και την καταπροτεραιότητα αποστολή ε, της ενέργειας. Εδώ είναι σαφές ότι για μορφές ενέργειας που δεν έχουν ε, διάρκεια στην ε, παροχή πρέπει να υπάρχει ε, πρόσβαση κατά προτεραιότητα. Πώς θα το δυσφαλίσω όμως αυτό αν θέλουμε να πετύχουμε το στόχο που έχουμε θέσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ξεπέρασα λίγο το χρόνο μου αλλά όχι όσο θα μπορούσα. ο πρόεδρος Μπούσεκ. Έχουμε εδώ τα ε, κόκκινα αστεράκια που βλέπετε στο χρονόμετρο. Ο κ. Κόχλιτσεκ τώρα, με συγχωρείτε, πολύ να ξεχάσω και συνάδελφε, από την Νοτική Αριστερά. Ευχαριστώ αγαπητέ πρόεδρε, μία ε, κατά βάση παρατήρηση από μένα. σχετικά με την αισιόδοξη ή υπεραισιόδοξη άποψη του φίλου μου Κλόντ που ξαφνιά φορά ξεχνά την πραγματική ζωή. Τα δίκτυα μας είναι της τάξης των 50 κύκλων. Και τι γίνεται και με τις γεωθερμικές αντλίες και με μεγάλα έργα ηλιακής ενέργειας όπως στην Ισπανία. Στην Ισπανία που χρησιμοποιούν κάτοπτρα. Τα κάτοπτρα διοχετεύουν την ηλιακή ενέργεια σε ένα ε, καυστήρα, ένα μποιλερ. εκεί ε, δημιουργείται ατμός κτλ. Πολύ ενδιαφέρον να τα δει κανείς αυτά τα πράγματα στο νότο της Ισπανίας όπου υπάρχουν. Θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και σε όλη την νότια Ευρώπη. Υπάρχουν και άλλα έργα που ανατρέπουν πολλά πράγματα. Όταν υπάρχει πολλή ενέργεια σε ένα σημείο, αυτό οδηγεί σε ανατροπές. Εγώ το λέω γιατί έχω και μία μικρή παραγωγή ηλιακών πάνελ. Όταν μιλούμε για την χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες ενέργειες, πρέπει να τα πούμε τα πράγματα αυτά. Πρέπει να τα λάβουμε υπόψη, ώστε να μην υπάρχει υπερσυγκέντρωση πόρων ανανεώσιμης ενέργειας σε ορισμένα σημεία όπου ενδέχεται να υπερεπιβαρύνουν τα δίκτυα στη Γερμανία εγώ συνιστώ να συνομιλήσετε με Γερμανούς συναδέλφους και διάφορους γερμανικούς φορείς καμιά φορά υπάρχει ο κίνδυνος blackout διότι το δίκτυο δεν αντέχει νομίζω ότι ο φίλος μου Κλοντ θα πρέπει να διαβάσει λίγα πράγματα αντί να αδιαφορεί. Και υπάρχουν και οι ιδιοσυλλεκτήρες σημαντικοί για την θέρμανση αλλά και για την προθέρμανση νερού που θα χρησιμοποιηθεί για άλλες χρήσεις εκτός από πόσιμο. Υπάρχουν τέτοιες χρήσεις σε ορισμένες ε, ευρωπαϊκές χώρες και τέτοιες εγκαταστάσεις. Όπως η χρήση της ε, θερμικής ενέργειας που ε, είναι υποπροϊόν παραγωγής άλλων ενεργειών. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί και αυτή η πηγή. Γιατί εγώ θέλω η έκθεση να είναι στο δυνατόν περιεκτικότερη όταν θα αναφέρεται στις διάφορες πηγές ενέργειας, χωρίς βεβαίως να αγνοήσει τους κινδύνους που διατρέχουν τα εφιστάμενα δίκτυά μας, διότι αν βελτιώνει κανείς κάτι χωρίς να ε, ε επεκτείνει και το δίκτυο, υπάρχει κίνδυνος. Άλλος κανείς? Κλοντ Τούρμες. Δεν σου φτάνουν τα 6 λεπτά. Τρία δευτερόλεπτα μόνο, Πρόεδρε. Θα σας στείλω μια πρόσφατη στατιστική από τη Γερμανία, απευθύνομαι στον Κόχλιτσεκ, που λέει ότι παρόλη την ελληνική ενέργεια έχει βελτιωθεί η ασφάλεια του γερμανικού δικτύου. Θα σου τη στείλω την επόμενη εβδομάδα. Και την επόμενη πέμπτη γίνεται μια διάσκεψη στις Ρυξέλλες από μια περιοχή της Γερμανίας που έχει την υψηλότερη ε, παραγωγή ενέργειας από ηλιακή ενέργεια κλπ. και θα είναι και ο υπεύθυνο εδώ. Ε, αυτό που έχει σημασία είναι η καινοτομία. Ευχαριστώ λέει ο ε, Μπούζεκ. Τώρα, εκ μέρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Ματίλντε Βάιστόρφερ, της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργεια, που είναι και διευθύντρια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και σα ευχαριστώ επίση κύριε Μπλάνκο Λόπες για την εξαιρετική έκθεση αλλά και την θαυμάσια συνεργασία που ε, μπορέσαμε να έχουμε μεταξύ των υπηρεσιών μας και του προσωπικού σας. Όλοι θεωρούμε ότι οι ανανεώσιμες θα πρέπει να παίξουν ηγετικό ρόλο, θα πρέπει να αυξηθούν, θα πρέπει να προωθηθούν και νομίζω και η έκθεση αλλά και ένα διτύπωσή μας της οδηγίας μαδίζουν στη σωστή κατεύθυνση. Και ασφαλώς, όπως είπαν και άλλοι συναδελφοί σας, θέλουμε να δημιουργήσουμε το πλαίσιο που θα επιτρέψει στους επενδυτές να έχουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Χρειαζόμαστε πολλούς επενδυτές στις ανανεώσιμες ενέργειες και πρέπει λοιπόν να είναι σωστό το πλαίσιο. Για παράδειγμα τώρα στην αναδιατύπωση σταματούμε οποιαδήποτε αναδρομικά μέτρα που έχουμε δει κάποιες φορές σε χώρες μέλη μας. Σαφές μήνυμα λοιπόν προς την αγορά και ευθυγραμμίζεται απολύτω και με τη Συμφωνία του Παρισιού. Θεωρούμε επίσης ότι η έκθεσή σας είναι καλή βάση για περαιτέρω συζητήσεις θα επανέλθω τώρα σε ορισμένα από τα σχόλια που έκαναν οι συναδελφοί σας κύριε Πρόεδρε και πρώτα για το στόχο. Θεωρούμε τον στόχο τουλάχιστον 27% δεσμευτικών μέτρων καλό στόχο και πάντως είναι ελάχιστο στόχος. Εάν επιτύχουμε περισσότερα τόσο το καλύτερο. Πάντως στη δική μας ανάλυση εμένουμε σε τουλάχιστον 27% δεσμευτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνδυασμό και με άλλα μέτρα του Clean Energy Package και ιδίω για την διακυβέρνηση όπου επίσης περιλαμβάνουμε προβλέψεις και για το ε, κενό των εκπομπών και για το gap filler. Όμως, πιο πολύ μας ενδιαφέρει ο στόχος. Περιλαμβάνει η της οδηγίας πολλά σχετικά στοιχεία. Μιλούμε για την οικονομική ανάπτυξη των ανανεωσίμων, όπως είπατε και εσείς, μειώνεται το κόστος των ανασύμων πηγών, ηλιακή, αιωλική κλπ. Ούτε καν η βιομηχανία δεν τα περίμενε αυτά πριν από έξι μήνες ή ένα χρόνο. Έχουμε λοιπόν εξαιρετικά θετικέ εξελίξει από την πλευρά του κόστου. Θέλουμε όμω να δώσουμε και περισσότερη δύναμη και στον καταναλωτή και αυτό συμπεριλαμβάνεται στην εκθεσή μα. Σε ό,τι αφορά την διεύρυνση τη αναδιατύπωση, μιλούμε όχι μόνο για το ηλεκτρικό ρεύμα, προωθούμε τη χρήση ανανεωσίμων ενεργειών και στην θέρμανση και ψήξη αλλά και στις μεταφορές. Και κάνουμε την πρόταση του 1% ανανεωσίμων σε θέρμανση ψήξη. Ο εισηγητής προτείνει 2%. Εμεί το θεωρούμε αυτό κάπως υπερβολικά υψηλό. Πάντως είναι σωστή η κατεύθυνση. Δηλαδή προώθηση περισσότερων ανανεώσιμων ενεργειών και στον τομέα θέρμανσης και ψήξη. Για τι μεταφορέ είχαμε και εξακολουθούμε και έχουμε στόχο. Θεωρούμε όμως ότι ο στόχος ίσως δεν απέδιδε σωστά. Γι' αυτό και δεν προτείνουμε στόχο τώρα, στην περίοδο μετά το 2020. Με την την να κλείσω το τηλέφωνο. Ο προηγούμενος στόχος ίσως δεν ήταν αρκετά διαφοροποιημένος και πάντως εν τέλει προωθεί κάποια βιολογικά καύσιμα βασιζόμενα σε καλλιέργειες, το οποίο δεν είναι αυτό που θέλουμε. Σε ό,τι αφορά το κόστος τεχνολογίας, προφανώς η αφετηρία μας υπήρξε προδιετίας όταν αρχίσαμε με το reference σενάριο και το policy σενάριο και όπως είπε και η Επίτροπός μας σήμερα το πρωί στον διαφρομένο διάλογο έχουμε αρχίσει ήδη να εξετάζουμε την ε, εξέλιξη του κόστους και συζητούμε νέους αριθμούς, νέα νούμερα και το σενάριο του κόστους για επίπεδα της τάξης 32-33% για να δούμε εάν θα υπάρχει διαφορετική, διαφορετικό αποτέλεσμα. Θα δούμε και οποιασδήποτε νέε μελέτες για τον τομέα αυτό. Γιατί είναι ταχύτατη εξέλιξη και ιδίως για το κόστος τεχνολογίας. Για αυτά που είπε ο Κλόντ για τη χρηματοδότηση, ασφαλώς είναι σημαντική η πτυχή αυτή. Και Κάποια δουλειά έχει γίνει ήδη και στο Ταμείο EFSI, το Ταμείο Juncker. Γίνονται βεβαίως και στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη που έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις και για την αποδοτική χρήση ενέργειας αλλά και για τις ανανεώσιμες. Οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε όπως πρότεινε ο πρώτη για τη διακυβέρνηση αλλά και για τις ανανεώσιμες συνολικότερα είναι καλή ιδέα και νομίζω θα ε, υποστηρίξουμε οτιδήποτε σχετική ενέργεια. Τέλο. Ένα θέμα που έθιξαν ορισμένοι συνάδελφοί σας, γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια σαφής διαίρεση έργου, κατανομή έργου που έχουν συμφωνήσει οι πρόεδροι των επιτροπών σας για τα διάφορα ε, σημεία, ε, για, την, ε, για τα κριτήρια της βιολογικής ενέργειας κλπ. Και αναμένουμε βέβαια και τη γνωμοδότηση της Ήτρα, όπως έκανε και η Επιτροπή σας ένβη περιβάλλοντος για τις άλλες πτυχές Είμαστε λοιπόν πολύ ανοιχτέ απέναντι σε αυτό το input. τέλο να πω ευχαριστώ στον εισηγητή και όλοι εισηγητάς και σε όλα τα υπόλοιπα μέλη σα, και πολύ ευχαριστώ να συνεχίσουμε την εργασία αυτή και οποιασδήποτε ερωτήσει έχετε ευχαριστώ να τις συζητήσουμε και ευχαριστώ και πάλι τον κύριο Μπλάνκο Λόπε. Ευχαριστώ. Σεις κύριε Σιγητά, είστε ικανοποιημένο κι εσεί. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θερμά ευχαριστώ σε όλους και θα ήθελα να πω στον συνάδελφο Κέλλη ότι η πράσινη γραβάτα μου, το χρώμα της Ισλανδίας, ε, την έβαλα επίτηδες για να καταφέρω να σας πείσω μέχρι τέλους. Γιατί θέλω να συμφωνήσετε κι εσείς με αυτούς τους στόχους που κατά βάθος ε, του εστεριζόμαστε όλου, που είναι να απεξαρτητοποιηθούμε από τον άνθρακα, να, απαλλαγούμε, να απαλλάξουμε την οικονομία μα από τον άνθρακα. Το θέμα δεν είναι ο στόχο, όλοι συμφωνούμε προ το στόχο. Ω προ το πότε θα τον υλοποιήσουμε ίσω διαφωνούμε. Αλλά νομίζω ότι έχουμε μια ιστορική ευκαιρία και μπορούμε να συμβάλλουμε και εμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να γράψουμε ιστορία με φιλόδοξου στόχου, Γιατί όλα, συμβαίν, όλα συμβαίνουν γύρω μα, το πρωί μα είπε ο κύριο Ζωρίνιο, ότι οι τελευταίες μέρες στις Βρυξέλλες ήταν από τις ε, μέρες τις πιο θερμές της ιστορίας. Θυμάστε τι έγινε τις προάλλες με τις πυρκαγιές στην Πορτογαλία. Όλα αυτά δείχνουν ότι κάτι έχει αλλάξει. Δεν μπορούμε εμείς ε, να θελοτυφλούμε ή να μένουμε με τα χέρια σταυρωμένα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Θα πρέπει να είμαστε διορατικοί και στις προτάσεις μας. Μερικοί στόχοι ε, της πρότασης υπολείπονται των ε, στόχων ε, του Παρισιού το, και οι μελέτες αντικτύπου πολλές φορές υστερούν σε σχέση με τα νέα στοιχεία. Επίσης, δεν θα πρέπει να απομονώνουμε αυτή την πρόταση. Έχουμε το στόχο μεγαλύτερης φιλοδοξίας. Είναι πολύ άριθμες οι μελέτες που υπάρχουν. Δεν ε, ήξερα αυτή τη ε, μελέτη της Ιρένα, αλλά έχω την ε, μελέτη του ΕΚΟΘΗΣ που λέει 35% χρειάζεται μερίδιο ΑΠΕ για να κρατήσουμε το βαθμό διείσδυσής τους της τωρινής δεκαετίας για την επόμενη δεκαετία. Αυτό λέει η μελέτη ΕΚΟΦΗΣ. Δεν ξέρω τη μελέτη Ιρένα αλλά έχουμε ως στόχο μεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά των ΑΠΕ. Επίσης, εθνικά δεσμευτικούς, εθνικούς δεσμευτικούς στόχους. Ξέρω ότι πολλές χώρες είναι κατά των δεσμευτικών στόχων. Αυτό όμως που έχει αποδείξει η υφισταμένη οδηγία είναι ότι Ακριβώς, αν θέλουμε να μιλούμε για μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ και αν σήμερα μιλούμε για μείωση του κόστου των ΑΠΕ, αυτό συνέβη ακριβώς γιατί στην ε, υφιστάμενη οδηγία οι στόχοι ήταν δεσμευτικοί για τις χώρες, γι' αυτό και λειτουργήσαν. Και γι' αυτό έπεσε το κόστος. Γιατί λοιπόν, αν κάτι λειτουργήσε τόσο καλά, εμείς να ομφαλοσκοπούμε αντί να κοιτούμε το παγκόσμιο συμφέρον, το συμφέρον για το περιβάλλον μας. Επιπλέον, η ασφάλεια δικαίου δίνει βεβαιότητα και σιγουριά στους επενδυτές και προσελκύει τις επενδύσεις για να επενδύσουν στην καινοτομία και να ρίξουν ακόμη περισσότερο το κόστος ε, των ΑΠΕ. Γιατί εκτό από βεβαιότητα θα δημιουργήσουμε πολλέ θέσει απασχόλησης και μάλιστα ποιοτική απασχόληση. Υπάρχουν λοιπόν πολλά αλληλένδετα και αλληλοσυμπληρώμενα σημεία. Φυσικά θα έχουμε και τομέακου στόχου. Μεγαλύτερη φιλοδοξία για απαλλαγή των μεταφορών από τον άνθρακα ή για τη θέρμανση, για την ψήξη και θα δούμε πώ θα τα υλοποιήσουμε όλα αυτά. Ε, και θα δούμε τι θα προτείνετε στι τροπολογίε σα. Πάντως θα πρέπει να συνεχίσουμε με τη μεγαλύτερη αποσαφήνιση και την ασφάλεια δικαίου και στους μηχανισμούς στήριξης. Επίσης θα πρέπει ε, να δώσουμε ενάψματα για την αυτοκατανάλωση, για να εμπλέξουμε και τους πολίτες, γιατί για πρώτη φορά μιλάμε για κάτι τέτοιο και θα μας βοηθήσει σίγουρα να υλοποιήσουμε το στόχο της απεξαρτοποίησης. Φυσικά σκεφτόμαστε και την Ιβηρική Χερσόνησο και την Ιρλανδία και άλλες περιοχές της Ευρώπης και γι' αυτό θα πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα των διασυνδέσεων, ώστε να έχουμε μια πραγματική ε, ενεργειακή ένωση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κάποια στιγμή θα πρέπει να γράψουμε ιστορία. Ας το κάνουμε από κοινού τώρα, ώστε να μπορούμε όλοι να συμμετέχουμε στην υλοποίηση στόχων που θα μας επιτρέψει μια ιστορική στιγμή να υψώσουμε μια ενιαία και ανεπιφύλακτη φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα διατρανώνει αυτούς τους στόχους. Εγώ Περιμένω πολλά από τη συνέχιση των εργασιών και το πνεύμα συνεργασίας που πριτάνευσε και στη σημερινή συζήτηση. Και επαναλαμβάνω και πάλι τις ευχαριστίες μου προς τη γραμματεία του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τους συνεργάτες, τους βοηθούς, ε, τους υπαλλήλους μας και μόνο με συνεργασία θα υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Μόνο με συνεργασία και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάποια στιγμή αργότερα στη διαπραγματεύση και με το Συμβούλιο. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπλάνκο Λόπες. Νομίζω ότι όλοι μείναμε ικανοποιημένοι και ευτυχείς. Λαμπρά. Η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών έχει οριστεί για τις 29 Ιουνίου 2017, δηλαδή έχετε μία εβδομάδα για να καταθέσετε τις τροπολογίες σας. Η επόμενη συνεδρίασή μας θα γίνει στις 10 και 11 Ιουλίου. Στις 10 και 11 Ιουλίου, τρεις μισές μέρες. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας και ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.